Uh, Φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλημέρα. Θα ξέρετε, ο κύριος Χέντελ επέστρεψε ως πρόεδρος της Επιτροπής. Υπέροχο, υπέροχη είδηση αυτή. Ήσασταν ο απόν φίλος μας και πιστεύαμε ότι θα επιστρέψετε στη θέση σας και τώρα επιστρέψατε και θα σας δώσω τώρα το σφυράκι και θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία και είναι καλό να ξεκινήσουμε από αυτό νομίζω ότι είναι απλή η ψηφοφορία παρακαλώ λοιπόν να συστηθείτε So, okay, Busmann. Hm? Micro. So, schönen guten Morgen allerseits. Ich will mich... Καλημέρα σε όλου. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για τι ευχέ σα. Όλε τι ευχέ κατά τη διάρκεια τη μακρά απουσία μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Με υποστηρίξατε. Πάρα πολύ. Και με βοήθησε πολύ η υποστήριξή σας και ευχές σας. Βλέπω ότι κάνατε πάρα πολύ δουλειά από ό,τι έμαθα πως με ενημέρωσαν σε διακομματικό επίπεδο. Αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να τακτοποιήσουμε κάποια πραγματάκια πριν ε, από το τέλος της ε, θητείας και σήμερα είναι ένα κομμάτι αυτού. Δεν έχουμε πολλά στην ημερήσια διάταξη, αλλά να τακτοποιήσουν κάποια θέματα. Ευχαριστώ και τη Μαρίτα όλο ιδιαίτερος, διότι η Μαρίτα ήταν ε, υπέροχη, αντιπρόεδρος, η οποία κάλυψε το κενό απουσία μου. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να γίνετε πρόεδρος. Έτσι της είπα, γίνετε πρόεδρος. Και αυτή είπε όχι. Όχι, μόνο, μόνο προσωρινά μέχρι να έρθετε. Κοιτάξτε, δεν είμαι 100% ε, έτοιμος ακόμα και δεν μπορώ να εργαστώ όπως συνήθως με 100% των δυνάμεών μου αλλά είμαι καθοδόν προς την ανάρρωση και την άκαμψη και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι αποτελεσματικό στην πρωί της Επιτροπής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις κανονικές εργασίες. Δεν έχει αλλάξει μέρη σε διάταξη. Οπότε εγκρίνεται. Δεν έχουμε μαλτέζικα, χροατικά, βουλγαρικά και ε, φινλανδικά ενεργητικά. Είναι μόνο παθητικά. Τώρα, πρακτικά της, της 23ης ε, ε, Ιανουαρίου. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ωραία. Εγκρίνονται. Περνάμε στο 4 που είναι η έκθεση η ο απολογισμός για τις διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Θα έπρεπε να πάρει το λόγο ο Γκυγιόν Μπελάς, δεν είναι όμως εδώ. Καλά, αυτό να βάλουμε τότε. Μετά τις ψηφοφορίες, μέχρι να επανέλθει. Για να μας ενημερώσει. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δεύτερο τμήμα για αυτό το σημείο. Ο συνάδελφος Λένας είναι εδώ και μπορεί να μας ενημερώσει για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και πάλι. Μπορώ να σας δώσω κάποια καλά μαντάτα όσον αφορά το θέμα. Την περασμένη πέμπτη το πρωί στο Στρασβούργο έγινε ο τελευταίος τριμερής διάλογος με τη Ρουμανική Προεδρία και τον Επίτροπο Τάισον ε, και καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας που θα ονομαστεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας και είναι σημαντικό το, βήμα αυτό για αυτή η ονομασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολύ καλά ισορροπημένη συμφωνία που λαμβάνει υπόψη πολλά σημαντικά στοιχεία που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθούν, όπως και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελεσματική παράγραφος που περιέχεται για κοινές, κοινούς ελέγχους και επιθεωρήσεις και κανόνες για διαμεσολάβηση μεταξύ κρατών μελών. Εν γέννη λοιπόν μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα και περιμένουμε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης την επόμενη εβδομάδα και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο επόμενο με τα χαράς να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, για να δούμε υπάρχουν ερωτήσεις. Στον συνάδελφο Λένας. Οκ. Okay. Δεν βλέπω. Α, παρακαλώ. Ο Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπον. Δύο πράγματα. Δεν μπορώ, Τομάς, να αντισταθώ, να εκφράσω, να εκφράσω την τεράστια ευχαρίστηση που σε βλέπω ξανά εδώ μπορούμε ξανά να συζητήσουμε, να τσακωθούμε. Αυτό μου έλειψε. Ο φάκελος του κυρίου Λένε είναι σημαντικότατος και τον συγχαίρω για τη δουλειά που έκανα. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος το λόγο παρατηρήσει ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Συνάδελφε όχι. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων σας. Ήμουν και ο συγκεκριτής με τον κύριο Λέναρ πρέπει να πω ότι συνεργαστήκαμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, συνεργαστήκαμε σαν άριστοι συνάδελφοι από ότι ο φόρο τιμής στον τρόπο διεξαγωγής των υπραγματεύσεων από τον κύριο Λέναρτς και οφείλεται στην επιδεξιότητά του ως διαπραγματευτή επιτυχία. Έχουμε πετύχει ε, πολύ καλά αποτελέσματα σε αφορά τη δικασία και την ουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες παρατηρήσεις. Ερωτήσεις. Η κυρία Χάκιν. Ευχαριστώ καταρχάς. Καλώς ήρθατε εκ νέου. Για να μην χρονοτριβώ και παίρνω το χρόνο της Επιτροπής, θα ήθελα να απηχήσω τα, αυτά που είπε και ο Σπάνης και όσον αφορά το συνάδελφό μας. Ωραία. Αλλά τώρα ήρθε ο, ο συνάδελφος Γκυγιόν Μπαλάς. Ας το αφήσουμε ένα λεπτό για να κάτσει και να ε, ξελαχανιάσει. Είμαστε στο 4-1 και αν μπορείς παρακαλώ. Από ό,τι κατάλαβα. Μου, μου τα είπαν λίγο σε κάτι άλλες γλώσσες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε τώρα και αυτό που σας ενδιαφέρει είναι οι επαναπτεύσεις για το 8.3. Να σας τα πω λοιπόν. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία είναι μάλλον δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί εάν δεν κλείσει η διαδικασία μέχρι, ας πούμε, στις αρχές Μαρτίου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε τελική συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό είναι προφανές. Γίνονται δύο παράλληλες συζητήσεις οι οποίες όμως γίνονται απλώς παράλληλα χωρίς να τέμνονται. Ε, δηλαδή, πρώτα έχουμε το θέμα του Κοινοβουλίου, το οποίο έχω την τιμή να εκπρόσωπω σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, εμείς επί όλων των σημαντικών θεμάτων έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει συμβιβαστικές προτάσεις σε σχέση με όλες τις τις αρχικές μας θέσεις, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποστοχωρήσει και όσον αφορά τον συνυπολογισμό και όσον αφορά το θέμα των διασυνοριακών εργαζομένων και όσον αφορά τις πολλαπλές δραστηριότητες. Ακόμα ε, και για θέματα εφαρμοστέας ε, συνολικής διαδικασίας εμείς έχουμε μετακινηθεί από τις θέσεις μας για να βρούμε πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σήμερα το Συμβούλιο που έχουμε απέναντί μας δεν θέλει να μετακινηθεί. Μετακινείται πολύ λίγο. Θεωρεί σε γενικές γραμμές ότι έχει μία θέση από την οποία δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω εσωτερικών ισορροπιών του Συμβουλίου και επομένως εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις θέσεις τους και στην πρότασή τους. Ωστόσο, μερικές από τις προτάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από πολιτικής απόψεως, αλλά και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή θα είναι πολύ επικίνδυνες εάν εφαρμοστούν. Ξέρω ότι εντωμεταξύ γίνονται πολλές συζητήσεις ε, γιατί ξέρω και μαθαίνω ότι γίνονται αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές εσωτερικές συζητήσεις στο Συμβούλιο. Ε, ο επόμενος τριμερής, μάλλον όχι, ε, η επόμενη συνάντηση των σκιωδών θα γίνει σήμερα το απόγευμα και ο επόμενος τριμερής αύριο. Θα δούμε τότε πού βρίσκεται η κατάσταση. Υπάρχει κάτι σημαντικό. Περιέργως ε, το ε, Συμβούλιο δεν θέλησε να γίνουν κάποια τριμερείς διάλογοι, αλλά αυτό δεν είναι η σωστή λύση αντιθετω Θα πρέπει να ε, έχουμε ακόμα περισσότερους τριμερείς αν θέλουμε να επιτύχουμε συμφωνία. Ε, βεβαίως υπάρχει και αυτή η ψυχολογική ένταση ε, ως ε, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί ξέρουν ότι απέναντί τους θα έχουν μια πολύ ε, δυνατή και ενωμένη ε, ομάδα κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και στους δύο κάθε επιτυχία στην περαιτέρω διαδικασία. Οπότε το Τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες. για τις προβλέψεις με συνθήκες εργασίας. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση. Είναι μόνο μία ψηφοφορία η οποία Πρέπει να είναι ονομαστική. Έχετε τις κάρτες σας όλοι, έτσι δεν είναι. Οπότε μπορείτε παρακαλώ να τις χρησιμοποιήσετε όπως πρέπει. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την πληροφορία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, 5 ε, κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. Η Μαρίτα θέλει να πει κάτι. Να πω μερικά λόγια. Εφόσον υποστήριζα τον κύριο Σαμπόν κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών συναντήσεων που έγιναν αργά το βράδυ πολλές φορές, θα του πω ότι ήταν καλό το αποτέλεσμα. Δεν ήμουν σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα τα καταφέρετε, αλλά ήσασταν τόσο αφοσιωμένο στην προσπάθειά σας που καταφέραμε να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα για όλα τα κράτη-μέλη. Και για μας που έχουμε αυτό το βόρειο, του σκανδιναβικό μοντέλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεκπαιρέωση αυτής της περιπλοκότατης εργασίας και για το καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ε, αν μου επιτρέπετε, σας ευχαριστώ τη γραμματεία, όλους τους συνεργάτες, όλους τους αδέλφους, ήταν πολύ σημαντικό το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των ε, συμπολιτών μας. Και από την πλευρά μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Οπότε, πάμε στο 6 το οποίο όμως θα αναβληθεί μέχρι την επόμενη φορά. Οπότε η επόμενη ψηφοφορία. προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες στην εργασία. Τρίτο τμήμα. Οπότε ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έχετε τις κάρτες σας, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Ψηφίσατε λοιπόν όλοι. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας. Και Πάμε ψηφί. Άριστα. Καταπληκτική εργασία. Ωραία. Οπότε, τελευταίο σημείο επί της ουσίας, το 8. Συζήτηση για το συντονισμό των ε, κοινωνικών ασφαλίσεων ε, να δώσουμε το λόγο στις εισηγήτριες Χάρκιν και Τζιν Λάμπερτ. Θέλετε παρακαλώ να παρουσιάσετε το θέμα. Η, η Μαρία Ευχαριστώ. Θα πούμε κάποια λόγια και δύο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ξέρετε, είναι πρόταση να έχουμε μέτρα ανάγκης στην περίπτωση του συντονισμού τη κοινωνικής ασφάλισης, στην περίπτωση ενός σκληρού Brexit, ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Πώς το προσεγγίσαμε. Το Κοινοβούλιο επέμεινε εξ αρχής ότι τα δικαιώματα των πολιτών έχουν την ύψιστη προτεραιότητα. Και όταν το συνδυάσαμε την ελευθερία μετακίνησης, έναν από τους τέσσερις πυλών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είδαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε σωστή λύση, να μην υπάρχουν κενά το δίχτυ ασφαλείας που δημιουργήσαμε να είναι επαρκές. Πολλές από τις άλλες προτάσεις όσον αφορά αυτά τα μέτρα ανάγκης υπερψηφίστηκαν χωρίς αλλαγές. Μικροαλλαγές υπήρξαν σε κάποιες προτάσεις μόνο. Αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, όπως σας είπα, επειδή έχει και αντίκτυπο στους πολίτες, και την ελευθερία διακίνησής τους πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικότατα το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Και θα πω κάτι που θα πούν και άλλοι. Το θέμα των υπηκών τρίτων χωρών. Το συζητήσαμε ήδη αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναντηθήκαμε με το Συμβούλιο και συνεδριάσαμε και σκιώδης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι είναι καλυμμένη βάσει του 1231, όχι του 883, προς διευκρίνηση. Να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα μπορούσε να μας διευκρινίσει την κατάσταση. Δηλαδή ότι οι πίκοοι τρίτων χωρών θα καλύπτονται είναι ερώτησή μου. Ε, έχουμε μέτρα ανάγκης για το 8, το 3, αλλά όχι για το 1231. Γιατί δεν χρειάζεται. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάλυψη. Παρόλο που το συζητήσαμε, θα είχαν την καλοσύνη να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μέτρου ή μέτρων όσον αφορά τους υπηκόους ε, τρίτων χωρών. Τα άλλα σχόλια αναφέρονται στις τροπολογίες που υποβάλαμε. Όπως τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δίποτε σχετικοί φορείς που θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα, είτε εθνική είτε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα έχουν επαρκείς πόρους. Διότι οι πολίτες θα θελήσουν απαντήσεις και μάλιστα γρήγορα. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες για τα χρονοδιαγράμματα και οι συνάδελφοι του γνωρίζω ότι έχουν κάποιε τροπολογίε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μία έκθεση σε ένα χρόνο. Θα προβαίνει σε μια αξιολόγηση του πώς λειτουργεί το όλο πλαίσιο και αν υπάρχουν πρακτικά θέματα ή προβλήματα. Υπάρχουν επίσης κάποιες τροπολογίες που αφορούν το ότι αυτή η νομοθεσία θεσπίζεται με την επιφύλαξη ή ενδήποτε διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών ή ενδήποτε μελλοντικών διμερών συμφωνιών ή συμβάσεων ε, μεταξύ κρατών μελών. Τέλος και τα υπόλοιπα υπόλοιπα θα τα αφήσω να τα πει η Τζιν. Θέλαμε οπωσδήποτε να υπάρξει κάποια δήλωση, μία αναφορά που θα αναφέρεται στη σημασία της αμοιβαιότητας, της καλής συνεργασίας, διότι ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί καλά αν συνεργάζονται ε, καλά τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι θετικό. Ευχαριστώ. Και η Τζιν Λάμπερ τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που αφορά τροπολογίες του ΕΛΚ. Εδώ. Αναφερόμαστε στις διμερείς συμφωνίες, ε, αλλά χωρίς ε, συγκεκριμένη αναφορά σε ενδεχόμενες μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρείτε ότι μπορούμε να βρούμε κάποια ε, διατύπωση η οποία ανακαλύπτει και το σημείο αυτό, ε, γιατί είχαμε και την έκθεση ας πούμε, το στο προηγούμενη θητεία ε, όπου έλεγε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει συμφωνίες και να προσπαθεί να κάνει συμφωνίες και με τρίτες χώρες. Βεβαίως κατανοούμε όλοι, όχι μόνο εγώ, ότι η πρόταση αφορά ε, σε αυτή τη, αφορά τη στιγμή ε, αυτή επίγοντα μέτρα ε, τα οποία πρέπει να ληφθούν, αλλά θα πρέπει ίσως να προβλέψουμε και κάτι που θα αφορά το μέλλον ε, και κάτι αντίστοιχο. Συμβαίνει και στο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται και αυτοί να μάθουν βέβαια τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μία φορά τουλάχιστον ας το κάνουν και αυτοί. Ξέρω ότι δεν το λέω με κινησμό, αλλά είναι πραγματικό γεγονός. Ε, έλεγα λοιπόν μήπως καταφέρουμε με κάποια διατύπωση να αφήσουμε και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να ευχαριστήσω μόνο τους συναδέλφους που δέχτηκαν να προσυπογράψουν και τις πρόσθετες τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρχεται η συζήτηση. Ποιο θα ήθελε να εκφραστεί? Ο Σβέν Σούλτσε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαι πρώτος που, που ε, μιλάει από πλευράς ε, του ΕΛΚ στη σημερινή ε, συνεδρίαση να σε ευχηθώ καλή ανάρρωση, ό,τι καλύτερο από πλευράς του ΕΛΚ και χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμη και αν δεν είστε ακόμη στο 100% σας εύχομαι να το ανακτήσετε τάχιστα. Τώρα για την έκθεση είμαι ο σκιώδης του ΕΛΚ Για μας ε, η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ταχύτητα και ε, η αποφασιστικότητα μεταξύ των εισηγητών. Αν προκύψει η ε, αποχώρηση χωρίς συμφωνία, που μπορεί να συμβεί, πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης που έχουν κάποια σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα βέβαια και τα δικαιώματα των πολιτών της ε, Βρετανίας στην Ένωση. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ε, ε, πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έλαβαν ιατρική βοήθεια και μετά δεν τους επιστρέφουν τα έξοδά τους και άτομα τα οποία έχουν εργαστεί για μεγάλο διάστημα στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα μπορούν να λάβουν την σύνταξή τους. Υπάρχουν γενικότερα θέματα Κοινωνική ασφάλισης. Και αν υπάρξει σκληρό Brexit, δεν θα είναι εύκολο να λάβουμε την αναγκαία προφόρηση και να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, γιατί θα είναι τρίτο κράτος η Ένωση. Πρέπει να υπάρχει περισσότερο νομική ασφάλεια, λοιπόν. Να δούμε πώς θα υπάρχει η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιαδήποτε αποχώρηση και αν υπάρξει πρέπει να την καλύψουμε. Οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Και αυτό υπόθηκε. Να καλύψουμε όλα τα ενδεχόμενα. Γιατί είναι δυνατόν ίσως να υπάρξει μια κυβέρνηση στον Ηνωμένο Βασίλειο η οποία κυβέρνηση να έχει ε, εχθρική στάση προς την Ένωση και να μην είναι διατεθειμένη να ανταλλάσσει στοιχεία με την Ένωση. Γι' αυτό, για μένα, θα είχε έννοια να σκεφτούμε ε, μήπως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη μεμονωμένα και διμερώς να συνάψουν συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί το βασικό θέμα για όλους τους πολίτες και τους δικούς μας και τους Βρετανούς το βασικό είναι η ταχύτητα των ε, ανταλλαγών προφοριών. Πρέπει λοιπόν ε, βεβαίως να παραμείνει ως plan ε, B αυτές οι διμερείς συμφωνίες. Η πρώτη μας λύση θα πρέπει να είναι να υπάρξει σωστή συμφωνία μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου. Αλλά αν δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία, τότε η ανταλλαγή προφοριών και δεδομένων που είναι απόλυτα αναγκαία πρέπει να είναι σίγουρη. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τώρα πολιτικές διακηρύξεις και να προσπαθούμε να κερδίσουμε μικροπολιτικά ωφέλη στην πλάτη των ε, ασθενών και πολιτών. Όπως είπα, αυτό θα ήταν ένα plan B. Μόνο εάν φτάσουμε στο σημείο που θα είναι δυσχερές να συνοηθούμε με το Λονδίνο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να συνοηθούν με το Λονδίνο επειδή το Λονδίνο δεν το επιθυμεί. Θα είχε λοιπόν έννοια τότε να υπάρξουν διμερεί συμφωνίε μεταξύ των κρατών μελών και του Λονδίνου απευθεία. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζουέν, Σούλτσε, ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Τόμας, χαίρομαι που επανήλθε. Χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Πολλοί σου ευχήθηκαν περαστικά, πολλοί εξέφρασαν την ε, αλληλεγγύη μαζί σου, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα παλέψει γιατί είσαι αγωνιστής και ξέρεις να παλέψεις. Τώρα για το περιεχόμενο. Το βασικό είναι ότι χρειάζεται ασφάλεια για τους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην τύχη τους. Δεν μπορούμε να πούμε είναι επισφαλής κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πρόσφατα. Συζήτησα με τους Πολωνούς που εργάζονται στην Βρετανία και μας είπαν ότι υπάρχει κυνήγι μαγισσών εδώ πέρα. Λέγεται να ξεκουμπιστούν όλοι οι Πολωνοί. Η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Και αυτό είναι σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η προσπάθεια ορισμένη να είναι έξαλλη κατά των Πολωνών. Πολλά υπόθηκαν και η Μάριον το είπε. Πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να επιδιώξουμε να υπάρξει διαρκής συνεργασία ε, αλλά δεν ξέρουμε πώς ε, θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ε, πιο σκληρή Και εμείς στη Γερμανία, στη, ως Γερμανοί πάντα επιχειρήσαμε να συμφωνήσουμε με τους Βρετανούς, αλλά το βασικό είναι ότι όταν συμφωνεί κανείς κάτι να τηρούν και οι δυο πλευρές τη συμφωνία. Βεβαίως προτιμούμε την ε, σύναψη ε, συμφωνίας με όλους, αλλά αλλιώς θα μπορούσαμε να έχουμε και διμέρες συμφωνίες. Κοιτάξτε, η κυρία Μέη μπορεί να πηγαίνει ως προσκυνήτρια σε διάφορα μέρη και να ζητάει διάφορες ειδικέ λύσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση. Η έξοδος αυτή δεν είναι δυνατόν να έχει σκληρότερε επιπτώσει ε, σε ορισμένε χώρε έναντι άλλων. Βεβαίω, πρέπει να είμαστε σαφεί, με πνεύμα συνεργασία, ούτω ώστε να φροντίσουμε, ούτω ώστε να υπάρχει ασφάλεια για του εργαζόμενου, ε, αν εργάζονται σε μια χώρα που στο μέλλον θα είναι τρίτη χώρα. Όταν θα ληφθεί απόφαση, δεν θα μπορεί να διορθωθεί μετά. Αλλά επίκυνται ε, εκλογές, όπως ξέρετε. Ε, εδώ ευρωεκλογέ. Και σε οποιαδήποτε εκλογή ε, είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν 52-48 σε αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε είναι πολύ μικρή διαφορά. Μπας, θα χάσουμε κάποιου καλού συναδέλφου. αλλά χαίρομαι μου που η Μάριον και η Τζιν ε, ήταν μαζί μας. Πάντα ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε και νομίζω ότι θα παραμείνει αυτό το κοινό πνεύμα οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπάρξει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, Τόμας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες. Με συγχωρείτε, ε, ξέχασα κάποιους σκιώδεις. Πρώτα απ' όλα ο Μπαλάς. Προς Θεού δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω ούτως ή άλλως. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και ξέρουμε ότι ο βαθμός προβλεψιμότητας ε, που μπορεί να έχουμε ε, και μετά και με από όλα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό δεν είναι ε, πολύ θετική. Έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες πολύ ενδιαφέρουσες αλλά παραμένει και ένα ερώτημα δηλαδή τι γίνεται με τους πολίτες πολίτες τρίτων χωρών. Αναφέρομαι σε πολίτες που ε, δεν ε, ε, προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα της συνέχειας των ανθρώπων αυτών είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες ε, προτάσεις, αλλά δεν ξέρω εν τέλει που έχουμε καταλήξει. Η Χέλγα Στίβενς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω μετά από είναι μακρά απουσία σας. Ε, καλή τύχη και καλή συνέχεια. Εγώ είμαι σκιώδης για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η κοινωνική ασφάλεια, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, αλλά προβληματίζονται οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στην ε, Μεγάλη Βρετανία, καθώς επίσης ε, προβληματίζονται και οι Βρετανοί, οι οποίοι ζουν εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστούν τα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλους αριθμούς. Είναι πολλοί ε, αυτοί οι οποίοι επίσης ζουν από τα ε, επιδόματα και τις ε, κοινωνικές παροχές και που δεν θα έχουν άλλη δυνατότητα επιβίωσης. Το θέμα βέβαια κατανοούμε ότι είναι περίπλοκο. Αυτό το δεχόμενο. Ε, εγώ λοιπόν θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες ε, γιατί έκαναν εξαιρετική δουλειά. Το έγγραφό τους είναι ε, μεγάλη υψηλής ποιότητος και βέβαια κανείς μας δεν θέλει αυτό το hard Brexit, αλλά εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τουλάχιστον πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα ε, συνεχίσουν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να βρούμε επικοδομητικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κατλίν Μπόιλεν. Α, καλά, δεν είναι εδώ. Η Ντανούτα Γιαζοβλέτσκα. Ευχαριστώ πολύ το μας. Σου εύχομαι εγκάρδια το καλωσορίσεις και πολύ πολύ υγεία. Σου εύχομαι. Και θέλουμε να είσαι παρόν στην επόμενη θητεία. Ο κανονισμός που συζητούμε θα, πρέπει να εξαλείψει αρνητικές συνέπειες του Brexit. Οι Βρετανοί και οι Ευρωπαίοι που, είναι εγκατεστημένοι στη Βρετανία διακατέχονται από βεβαιότητες όσον αφορά το μέλλον τους. Έχω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζομένους και τους πολίτες τρίτων χωρών. Έθεσα ερωτήσεις όσον αφορά την κατάστασή τους. Σαν απάντηση έλαβα τη διαβεβαίωση το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ τους εισηγητές, ε, τους κοιόδης για την εργασία τους. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς των εισφορών σε χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Θα πρέπει να προβλέπετε μια λύση στον κανονισμό. Θα πρέπει Πρέπει να αναλύσουμε τις διάφορες προτάσεις, τις προτάσεις του συναδέλφου Σούλτσε ε, λεπτομερώς, διότι παρέχονται κάποια χέγγια, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να εφαρμόσουμε αυτές τις προτάσεις σε διάφορες καταστάσεις να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ασφάλιση και στους Βρετανούς και στους πολίτες των τρίτων χώρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Άλλος. Κανείς. Οπότε, οπότε ο Ζόρντι Κουρέλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δύο είδη ερωτήσεων έχουμε. Καταρχάς, όσον αφορά την κάλυψη παρέχει αυτή η πρόταση σε προσωπικό επίπεδο και μετά υπάρχουν και οι ερωτήσεις για του προστασμένους εργαζομένους και τι υπηκότητε των χωρών. Για του προστασμένους εργαζομένους αυτό που θα συμβεί τη στιγμή τη απόσυνομενου του Ηνωμένου Βασιλείου αν δεν υπάρχει συμφωνία είναι ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή, Ενώσεω θα πάψει και αποσπασμένοι εργαζόμενοι εργάζονται σε άλλη χώρα μόνο στα πλαίσια της αποσπάσεως. Αυτοί οι άνθρωποι, οι εταιρείε μάλλον, δεν θα μπορούν να εργάζονται στην Ευρώπη. Για το πρώτο 24 οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι όταν έχουν αποσπαστεί σε άλλο κράτο μέλο εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορέ στο κράτο μέλο καταγωγή του. Δηλαδή αυτοί που είναι ασφαλισμένοι στον Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται για μια εταιρεία βρετανική που παρέχει υπηρεσία σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το πρώτο 24 μήνο αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν εισφορέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα μετά την απόσταση. Μετά από το 24 μήνο αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώνουν εισφορέ στη χώρα στην οποία διαμένουν. και θα καλύπτω την πρόταση οδηγίας. Και θα ισχύουν τα εχέγγυα για το συνυπολογισμό, για ισότιμη αντιμετώπιση κλπ. Αυτό για τις χωρών είναι διαφορετική.